πρώτη είναι η έκθεση του κυρίου ε, Φάρια για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών. Κύριε Φαρία, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ε, συνάδελφοι, οι ωκεανοί και οι θάλασσε καλύπτουν το 70% τη επιφάνεια του πλανήτη και το θαλασσινό νερό αντιστοιχεί στο 97% των υδάτων του. Έχουν, παρέχουν τροφή, ενέργεια, κινητικότητα, θεραπεία και αναψυχή, ρυθμίζουν το κλίμα κλπ. Ε, οι ωκεανοί με τι παράκτιου και θαλάσσιου πόρου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, ε, οι οικονομικοί κλάδοι που αντιστοιχούν στους ωκεανούς αντιστοιχούν στο, στα 3,4 ε, ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, οι, οι, οι αντίστοιχες οικονομίες ε, εξαρτώνται πάρα πολύ από την βιωσιμότητα. Επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην, ε, στις αλλαγές του κλίματος, απορροφώντας περίπου το 25% των, του διοξιδίου του άνθρακα, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ε, βοηθώντας την αύξηση του οξυγόνου. Γι' αυτό το λόγο συμπεριλήφθηκαν στην Συμφωνία του Παρισιού. Ε, Όμω, ε, οι ωκεανοί και οι θάλασσε επηρεάζονται πάρα πολύ από τα κλιματολογικά φαινόμενα και είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η ισορροπία του. Ε, η μόλυνση και η μείωση της βιοπικιλότητας τα απειλούν. ο πληθυσμός της γης θα φτάσει ενδεχομένως στα 9 δισεκατομμύρια το 2050 και αυτό θα αποτελέσει μια πρόσθετη πίεση στις θάλασσες. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα χρειάζεται καλύτερη διεθνής διακυβέρνηση ε, και ενίσχυση των προσπαθειών σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό αναγνωρίστηκε και στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη ε, που καθόρισε ως στόχο την διατήρηση των ωκεανός. Είναι, ωκεανών. Είναι ένας από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Κομισιόν, ε, ή μάλλον η, η, η, η Κοινή Ανακοίνωση Επιτροπής και είπα του εκπροσώπου ε, αποτελεί τμήμα της απάντησης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και βασίστηκε σε μια ευρεία συνένεση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την διακυβέρνηση των ωκεανών, να μειώσουμε τις πιέσεις που δέχονται αυτοί και γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη γνώση των ωκεανών και των θαλασσών. Γι' αυτό το λόγο εγκρίθηκαν 50 δράσεις ε, προκειμένου οι ωκεανοί να αναπτυχθούν με τρόπο βιώσιμο. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάπτυξη και η ε, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή είναι οι τρεις άξονες στις οποίες θα πρέπει να κινηθούμε. Οι ωκεανοί βρίσκονται σε όλο και πιο ανησυχητική κατάσταση, γι' αυτό το λόγο επίγει να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να δράσουμε όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. Η έκθεση που θα ψηφιστεί αύριο δίνει την Κομισιόν να αναπτύξει εταιρικέ σχέσεις ε, με τους ε, βασικούς φορείς στον τομέα των ωκεανών ως μέσο για την επίτευξη καλύτερης διεθνούς διακυβέρνησης ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Επίτροπος κ. Βέλα το ανέφερε στη διάσκεψη για τους ωκεανούς. Είπε ότι οι ωκεανοί είναι η καρδιά της γης και εμείς θα πρέπει να τους διατηρήσουμε ζωντανούς. Αυτό είναι το καθήκον μας. Θα πρέπει να τους προασπίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύστημα παγκόσμιου συντονισμού των προσπαθειών μας. Ε, Ελπίζω ότι θα υπερψηφίσετε αυτή την έκθεση αύριο. Ευχαριστώ. Περνάμε κατευθείαν στο Catch the Eye. Κυρία Πιτικάιν, για ένα λεπτό. First of all, I would like to... Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φάρια για την εξαιρετική του έκθεση. Θα ήθελα να επανεπισημάνω κάτι που έχω πει και προηγουμένως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πρωτοστατήσει για μια ε, καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών ε, και μια ε, διεθνώς δεσμευτική σύμβαση που θα καλύπτει διάφορους τομείς που θα, θα καλύπτει την υπεραλίευση συγκεκριμένων αποθεμάτων ικθείων, ε, τις περιοχές ε, διατήρησης των ειδών ε, και τις, ανά, δράσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η οξύνηση των υδάτων και η, την ύπαρξη χημικών στα θαλάσσια ύδατα, όπως επίσης και στο πλαίσιο των αρχών της πρόληψης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης και τα μικροπληκτικά πλαστικά που είναι ε, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που υπάρχουν. Ε, σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία για το μέλλον, καλή επιτυχία και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θα αρχίσουν οι διαδικασίες ε, το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έξτρομ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κύριο για την πολύ καλή συνεργασία και για την πολύ καλή έκθεση. Πραγματικά είναι πάρα πολλές ε, οι ε, προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ε, ο πλανήτη και ιδίως σε ό,τι αφορά του ωκεανούς. Οι αλληλευτικές επιχειρήσεις σίγουρα και οι δραστηριότητες έχουν μεγάλη ευθύνη, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες δραστηριότητες που επηρεάζουν, όπως παραδείγματος χάρη η εξόριξη στα βαθαία ύδατα για ανέβρεση πετρελαίου, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Θα πρέπει να δούμε τι αποφάσεις ε, λήφθησαν σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις πετρελαίου ε, σε βαθέδατα. Πιστεύω ότι στο μέλλον ε, θα πρέπει να μπορούμε τις γενιές τις επόμενες να, ε, να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον υγιές και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να βοηθήσουν. Ευχαριστώ. Virkkunen. Arvoisa Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο κύριο Φάρια για αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Ξέρουμε ότι η μόλιση των ωκεανών είναι μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα τα πλαστικά. Το 95% των πλαστικών στον κόσμο χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και μετά τα πετάμε στα σκουπίδια. Και τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν στους ωκεανούς των ωκεανών απορρίπτονται στα νερά κυρίως πλαστικές σακούλες και πλαστικά μπουκάλια. Θα πρέπει να εργαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ καλό που οι πλαστικές σακούλες πλέον στην Ευρώπη χρεώνονται ε, και ανακυκλώνουμε τα πλαστικά μπουκάλια σε μεγάλο βαθμό στη Φινλανδία. Εδώ και δεκαετίες δίνουμε το καλό παράδειγμα ανακυκλώνοντας πλαστικά μπουκάλια. Το 92% των πλαστικών μπουκαλιών που πολλούνται ανακυκλώνονται στη χώρα μου. Αυτό θα πρέπει να γίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ε, ένα άλλο βήμα θα πρέπει να είναι η απαγόρευση των μικροπλαστικών. Η στρατηγική της ε, Χρειάζεται μια στρατηγική της Κομισιόν για το πλαστικό. Ευχαριστώ. Πολτσεκ. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Η κρίση που ζούμε στους ωκεανούς και στις θάλασσες ε, είναι τεράστια. Το, ο στόχος 14 του, της ε, ε, ατζέντας του για τη βιώσιμη ανάπτυξη μας υπαγορεύει να προστατεύουμε τους ωκεανούς. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική για τη βιοπικιλότητα αλλά και για τη ζωή των ανθρώπων στο περιοδικό Science δημοσιεύθηκε ένα άρθρο το οποίο κάνει λόγο για το πώς μπορούμε ήδη να εντοπίσουμε νεκρές ζώνες στους ωκεανούς και στις θάλασσες. Ανοιχνεύονται νεκρές ζώνες. Νεκροί υδάτινοι όγκοι. Πρέπει να συνεργαστούμε σε διεθνές επίπεδο ε, ε, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη γεωργία, για παράδειγμα τις θαλάσσιες μεταφορές. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Κύριε Έτμαν, θέλετε να συμμετέχετε στο Catch Λίγο πιο νωρί να μας το λέτε, γιατί πρέπει να οργανώσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε το λόγο και μετά θα πάρει το λόγο ο Επίτροπος Βέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη που με ανοιχτήκατε, δεν μπόρεσα προηγουμένως, άργησα να ε, δηλώσω ότι ήθελα να συμμετέχω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη διακυβέρνηση των ωκεανών, όχι μόνο γιατί έχουμε ευθύνε όσον αφορά του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί, δεν μπορεί κανένα άλλο μέρο στον κόσμο και θέλει από πλευρά μα μια πολύ σαφή ηγετική προσέγγιση. Έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια στην ανακύκλωση, όμω στην ανάπτυξη αγορών άλλων μερών ε, στον κόσμο. Αν αυτέ ε, οι αγορέ ε, δεν υπάρχουν στο μέλλον, μέλλον, αυτό, στο μέλλον αυτό δεν θα έπρεπε να ε, μειώνει τη δική μας δέσμευση να ε, συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν το κάνουμε εμείς, κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις θάλασσές μας, στον τομέα της επαγγελματικής αλίας, των πλαστικών, όλο αυτό το ζήτημα της ε, ρήπανσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ηγετική στον τομέα αυτών και γι' αυτό ακριβώ είναι μεγάλε οι προκλήσει μπροστά μα μεταξύ των 28 μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε να πρωτοστατήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριο Βέλα για να συνοψίσει την συζήτησή μα. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Φάρη και τον κύριο Μοντέλο Ντελβιλάρ όπως επίσης και τους κοιόδης εισηγητές ε, για την χρήσιμη και πολύτιμη δουλειά τους. Ε, εγώ επικροτώ την έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διακυβέρνηση των ωκεανών σε διεθνές επίπεδο και συμφωνώ με τους γενικούς στόχους της κοινή ανακοίνωση και των δράσεών τη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ για τα χρήσιμα σχόλιά τους. Αυτή η κοινή ανακοίνωση είναι ένα μεγάλο βήμα προς, τα μπρος. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ Εκπρόσωπο ε, ε, κάνει μια τέτοια δήλωση σε σχέση με τη διακυβέρνηση των ωκεανών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι πρωτο, πρωτοστατεί για την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. Η επιτυχής ε, έκβαση τη της σχετικής διάσκεψης στη Μάλτα πριν από μερικούς μήνες ε, δείχνει ότι είμαστε στην πρώτη θέση όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκοσμίων ε, προκλήσεων. Ε, το θέμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της ανταπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ε, το στοιχείο 23 ε, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με συγκεκριμένες δράσεις για τρεις τομείς προτεραιότητας για ασφαλέ, ασφαλείς, καθαρούς και βιώσιμα διαχειριζόμενους ωκεανούς. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο χρειάζεται ε, ένας ε, πιο συνολικός τρόπος ε, διακυβέρνησης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες σε διεθνές επίπεδο, όμως δεν υπάρχει πραγματική παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς, μια, χωρίς, χωρίς συγκεκριμένα κείμενα. Γι' αυτό εμείς ενισχύ, ενισχύουμε σε πολυμερές επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και σε διμερές επίπεδο και σε συγκεκριμένα προγράμματα την προσπάθεια αυτή. Προς αυτή την κατεύθυνση ενίσχυση του του, της, της, του του, της πολυμερούς προσέγγισης για τα θαλάσσια θέματα είναι πάρα πολύ σημαντική για να υπάρχουν προστατευμένες ασφαλείς θάλασσες, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συνεργατικών προσπαθειών. Γι' αυτό ακριβώς επικροτώ όλος ιδιαίτερος την απόφαση την περασμένο μήνα από, τη, από την ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να υπάρχει μια διεθνή συνέλευση για την επεξεργασία ενός κειμένου, ενός διεθνούς, διεθνώς δεσμευτικού ε, κειμένου από την UNCLOS για την θαλάσσια βιοπικιλότητα πέραν από κάθε εθνική δικαιοδοσία, γιατί σε αυτό είχε πρωτοστατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά χρόνια. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ε, μειώσουμε τις πιέσεις ε, στους ωκεανούς πιέσεις ε, και αιτίες προβλημάτων ε, που προέρχονται από τα θαλάσσια απόβλητα, ε, τη θέρμανση των ωκεανών, η οξύνηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών και της βιοπικιλότητας. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητες. Επίσης, εξαρτάται και από το σωστό προγραμματισμό και τη διαχείριση της ανθρώπινης χρήσης, ενθάρρυνση καλύτερης χρήσης θαλάσσιας χωροταξίας και καλύτερη διαχείριση και σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο. Και χαίρομαι όλο ιδιαίτερος που, που βλέπω ότι υπάρχει η υποστήριξή σας ως προς αυτό. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική για τα πλαστικά, αυτό θα συμπληρώσει τον αγώνα μας κατά ε, των θαλάσσιων απορριμμάτων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια για αναπτυσσόμενες χώρε ω ενδεχόμενη πηγή ε, τροφίμων, ε, θέσεων εργασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει βιώσιμη αλία, θα, ε, θαλάσσιες περιοχές προστατευόμενες, ε, μετριασμός ε, των ε, κλιματικών αλλαγών και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την θαλάσσια ασφάλεια. 590 εκατομμύρια ευρώ και ενδεχομένως ακόμη περισσότερα ε, προβλέπονται ε, στο πλαίσιο του, της περίοδου 2014-2020. Επίσης θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τους ωκεανούς, επομένως θα επενδύσουμε σε πάνω, πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ε, σε προγράμματα θαλάσσιων ερευνών, γιατί έχουμε νέες τεχνολογίες που ανοίγουν νέες δυνατότητες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε καταλήλως. Κάτι ακόμη, ένας ακόμη στόχος είναι να διερευνήσουμε περισσότερο τους ωκεανούς και να υπάρχει ένα δίκτυο θαλασσίων δεδομένων ανοιχτό σε όλους. Θα ε, υπάρξει επίσης ε, ε, συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο και κάθε δράση που έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση του ωκεανού ή με την πίεση προς το θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια ασφάλεια και την έρευνα όλα αυτά είναι τμήμα μιας σφαιρικής προσέγγισης. Υπάρχει μια λογική στο πλαίσιο αυτή τη προσέγγιση. Η πίεση προ του ωκεανού δεν είναι μόνο παγκόσμιο ζήτημα, αλλά ε, συνδέονται ε, μεταξύ τους τα διάφορα προβλήματα όπως και οι λύσει. Δεν εξαρτάται η επίλυση του προβλήματος μόνο από εμά, αλλά και από τους διεθνείς εταίρους μας και γι' αυτό το λόγο η υποστήριξή σα ε, για την δημιουργία σχέσεων συνεργασία για του ωκεανού είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα στη δυνατότητα να εντοπιστούν θέματα κοινού ε, συμφέροντος ε, και νέα ζητήματα για τους ωκεανούς. Ε, σας ευχαριστώ πολύ.